El Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Κυρίσω την έναρξη της συνεδριάσεως και ως πρώτο σημείο προβλέπεται η έκθεση του κυρίου Κάλφιν για τη χορήγηση εγγύηση Ευρωπαϊκής Ένωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσει για σχέδια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δώσουμε ευθύ αμέσω το λόγο στον κύριο Κάλφιν. Κύριε Κάλφιν, γνωρίζετε πως έχετε τέσσερα λεπτά στη διάθεσή σας προβλέπονταν έξι, αλλά δύο θα σας δοθούν για, στο κλείσιμο της συζήτησης. Τώρα, εάν θέλετε να μιλήσετε έξι λεπτά τώρα στην εισαγωγή, εντάξει, δεν θα έχετε στο τέλος χρόνο να μιλήσετε. Για άλλους τέσσερα συν δύο στο τέλος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, η παρούσα εντολή τη Ευρωπαϊκή Τάξη Απενδύσεων για τι επιχειρήσει εκτό Ευρωπαϊκή Ενώσεω εκπνέει τέλο Οκτωβρίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν επί των συνθήκων και των όρων για την παράταση τη